Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Την ημερήσια διάταξη την έχετε λάβει, δεν πιστεύω να χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχετε κάποιο έτοιμο για αλλαγή, όχι. Δεν έχω καμία ανακοίνωση να κάνω και εγώ, οπότε περνάμε κατευθείαν στο σημείο 3. Ενδιάμεση αξιολόγηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιφορική πλοήγησης, υλοποίηση, μελλοντικέ προκλήσει και προοπτικές χρηματοδότησης. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει μια νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας ε, του κύριου Ρέμεκ, τον οποίον ορίζω είναι ο υπεύθυνο και μας ε, παρακάλεσε σήμερα να κάνουμε μία μικρή ακρόαση μια μισή ώρας. Καλώς Καλωσορίζω λοιπον κάποιους εμπειρογνώμονες, τον κύριο Αλέν Μπένετο, την κυρία Μπάζη Πατάκη, η οποία ήταν μέλος της ε, Επιτροπής μας, τον κύριο Ζανζακ Τορτόρα, και τον κύριο Τόμα Στάρεκ. Έχουμε προσκαλέσει αυτούς τους ειδικού και σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι για να μας δώσουν ε, πληροφορίες. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση δημόσια που είναι απαραίτητη για να δούμε και βεβαίως να δούμε και κριτικά το μέλλον αυτού του έργου. Νομίζω είναι όλοι παρόντες, οπότε μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε ότι μπορώ να δώσω τον λόγο και να σταματήσω μιλάω και πρώτα απ' όλα στον κύριο Μπενετό που βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Κύριε Μπενετό, έχετε τον λόγο. Να σας υπενθυμίσω να προσπαθήσετε στον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων να ολοκληρώσετε εντός 10 λεπτών γιατί έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις οι ε, συνάδελφοι και εσείς να απαντήσετε πιο αναλυτικά. Αυτά αρκετά νομίζω με τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, κύριε Μπενετό, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και τον εισηγητή σας, τον εισηγητή της Επιτροπής ε, Ήτρε για τα θέματα του Γαλιλαίου που με προσκάλεσε. Δεν είμαι ποτέ μέλος Επιτροπής σας, αλλά προσεκλήθη ως πρόεδρος ενός ε, νεοπαγούς δικτύου που ε, υπάρχει εδώ και ένα χρόνο. Είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειών που χρησιμοποιούν ε, τις τεχνολογίες του διαστήματος. Πρόκειται για το δίκτυο Νερέους. Απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 26 περιοχές, περιφέρειες, 12 κρατών μελών. Ο στόχος του δικτύου νερέους είναι απλούστατος. Προωθεί μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των περιφερειών, γιατί οι περιφέρειες είναι καταλληλότερες για να πειραματιστούμε τις εφαρμογές και τροφοδοτούν μια ροή πληροφοριών ανάμεσά τους και ανάμεσα στις περιφέρειες και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις. Στόχος λοιπόν του Νεραίους είναι ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος με δύο μεγάλα προγράμματα, το GPS και το πρόγραμμα Γαλιλαίο, το GNSS. Γιατί αυτά τα δύο προγράμματα περιλαμβάνουν όλες τις εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης. Από τις ανταλλαγές απόψεων του δικτύου καταλήξαμε σε μία ομάδα εργασίας που ήδη συνεκλήθη, όπως σας είπα το δίκτυο είναι νεοπαγές Ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο, οπότε δεν έχει πλούσιο έργο ακόμη να επιδείξει. Αλλά από διάφορες ανταλλαγέ απόψεων που έγιναν για θέματα δορυφορικής πλοήγης καταλήξαμε στη σύσταση ενός γκρουπ εργασία, ε, μιας ομάδας εργασία που συνεδριάζει τακτικά και προωθεί μια ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια μια συμφωνία με την GSA Γαλιλαίο και Βλέπουμε πώς αναπτύσσονται οι διάφορες εφαρμογές και πώς συμβάλλουν εκεί οι περιφέρειες και τα κοινοτικά όργανα. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ε, κάποιος Ιταλός από την, από την περιφέρεια Βενέτσι. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ συχνά για τις εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης, αλλά και για άλλα προγράμματα, μιλούμε για τη δημιουργία πόλων αριστείας, clusters, για συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημιακών κύκλων, πανεπιστημίων και διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο αυτό υπάρχει μία ανοιχτή συζήτηση. Ποιοι κλάδοι είναι καταλληλότεροι για την ε, εφαρμογή αυτών των ε, προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης. Είναι οι μεγάλες ε, εταιρείε που εκπροσωπούνται στου πόλου αριστείας και ανταγωνιστικότητα, ή μήπω είναι καλύτερα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει καταλληλότερε για τι εφαρμογές αυτέ. Και εκεί δυστυχώ υπάρχει διάσταση απόψεων και διαφωνία. Για το δίκτυο νερέως που, που εκπροσωπώ εγώ εδώ σήμερα, είναι προφανέ ότι και ο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ζωτικό και θα πρέπει να προωθηθεί και να αξιοποιηθεί. Πριν από λίγο αναφέρθηκα στην ομάδα εργασίας ε, Πεγκάς, Πίγασος, ε, της Τζέσα Γαλιλαίο, που επεξεργάζεται μια πολύ σημαντική πρόταση που υποβάλαμε. Ζητήσαμε από τη ΖΕΣΑ Γαλιλαίο να βοηθήσει για, για την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου και σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε διαπεριφερειακό επίπεδο προκειμένου να καταρτιστεί ένα σαφής απολογισμός του βιομηχανικού ιστού που μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες εφαρμογές δορυφορικής υπολογής και να τις αναπτύξει αλλά να γίνει και μια εξαντλητική χαρτογράφηση των πεδίων εφαρμογής που είναι πολλά και διάφορα και έχουν εγκάρσιο χαρακτήρα. Πολύ συχνά, σε πολλές περιπτώσεις, ίσως είναι πιο σημαντικό να αναπτύξουμε τέτοιες κατακόρυφες δομές ε, και τέτοια αμοιβαία συνεργασία, αντί να αναζητήσουμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες. Γιατί υπάρχουν ε, σημαντικά περιθώρια πρόοδου με, την, ε, με το πλησίασμα κάποιων παραγόντων που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την αμοιβαία προσέγγιση. Μεταφορές, υγεία, γεωργία είναι τομείς που μπορούν να υποφεληθούν από αυτές, από αυτές τις εφαρμογές και στη Γεωργία υπάρχουν ε, τεράστια προβλήματα άρδευση, για παράδειγμα. Οπότε οι εφαρμογέ δορυφορική πλοήγηση είναι σημαντικέ και για του κλάδου αυτού. Δεν υπάρχουν τέτοια παρατηρητήρια και υπάρχει πολύ λυπή γνώση και εντό των περιφερειών και μεταξύ των περιφερειών, αλλά και μεταξύ περιφερειών και κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Η ομάδα εργασία ε, του Νερέους για τις εφαρμογές της δορυφορικής πλοήγησης εκπώνησε ένα εγγραφό που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και που κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον και σημαντικό έγγραφο και θα αναφέρω τρεις από τις προτάσεις του εγγράφου αυτού που κατά τη γνώμη μου χρήζουν επισήμανσης. Η πρώτη πρόταση είναι ότι στις περιφέρειες χρειαζόμαστε μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ε, ανάπτυξη και την εξέλιξη του προγράμματος Γαλιλαίο. Δεν θα σας κάνω μια ιστορική επισκόπηση της ε, ίδρυσης ε, του Γαλιλαίου, αλλά είναι προφανές ότι στις περιφέρειες και για την εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρειάζονται κάποια εχέγγυα για το μέλλον σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του προγράμματος Γαλιλαίος. Η δεύτερη παρατήρηση του εγγράφου αφορά τη χρηματοδότηση των εφαρμογών ε, και την ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής πλοήγησης. Είχαμε το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και, εκεί προβλέπεται χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και εκεί απαιτούνται ανταλλαγές για τη δυνατότητα αμοιβές αξιοποίησης αυτών των ε, κονδυλίων και να κρατήσουμε μια συνέπεια και συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση των κονδυλίων αυτών. Συνδυάζοντα τα κονδύλια του 7ου Ερευνητικού Προγράμματο Πλαισίου και τα κονδύλια του Ταμείου Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή. Το περίφημο Ταμείο ΦΕΝΤΕΡ που για την επόμενη δεκαετία θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτηση. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια του ΦΕΝΤΕΡ. Είναι σημαντικά ποσά που θα συμπληρώσουν ε, τα κονδύλια του 7ου Ερευνητικού Προγράμματος Πλαισίου. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε στη συζήτηση. Και τρίτο θέμα που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας για το GNSS Νερέους είναι η ανάγκη διάδοσης ε, της πληροφορίας και της γνώσης. Μπορεί να σας εκπλήξω, αλλά εκεί που αναπτύσσονται οι εφαρμογές, δεν υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, αρκετοί φορείς που να έχουν γνώση εμπεριστατωμένη και να μπορούν να χειρίζονται καλά τις δυνατότητες του Γαλιλαίου. Πολύ συχνά έχουμε κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινητοποιούνται στο θέμα αυτό, αλλά σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης υπάρχουν κενά πληροφόρησης και επικοινωνίας. Και εκεί το δίκτυό μας, το δίκτυο Νερέους, ζητά επίμονα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα μια βελτίωση της επικοινωνίας, μια καλύτερη διάδοση και προβολή των διαφόρων εφαρμογών του προγράμματος Γαλιλαίο. Γιατί υπάρχει λυπή ενημέρωση, όπως σα είπα. Και αυτό το κενό θα πρέπει να το καλύψουμε. Ένα άλλο σημείο, γιατί μιλούμε για το Γαλιλαίο μαζί με το έγνος Πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι στη δική μου περιοχή, περιφέρεια, Μιντι Πυρενέ, πολύ λίγοι γνωρίζουν για την συνέργεια Γαλιλαίο Έγνος. Και ακόμη και σε εταιρικέ σχέσεις που είχαμε με την περιφέρεια της Μαδρίτης, ε, ελάχιστοι γνωρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες αυτής της συνέργειας. Μιλούμε πολύ για το έγνος και για την πιστοποίηση του σήματο έγνος. Το γεγονό ότι το σήμα έγνος ε, θα κρυθεί κατάλληλο για την ε, αεροπορία είναι πολύ σημαντικό για τις εφαρμογές και το γεγονό ότι η πολιτική αεροπορία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μήνυμα θα είναι σημαντικό, αυτό το σήμα μάλλον. Και μια και μιλάω για επικοινωνία, θα ήθελα να εκφράσω εδώ την ε, επίμονη ανάγκη επικοινωνίας για το τι εστί το σήμα έγνος σε σχέση με το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Σήμερα οι συμπολίτε μου γνωρίζουν το GPS, το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, άκουσαν κάτι ψηλά για το Γαλιλαίο. Η σχέση όμως Γαλιλαίο-Έγνο και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής είναι κάτι που μένει πολύ γενικό και αόριστο για τους περισσότερους. Θα σα δώσω μερικά παραδείγματα, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο για τις περαιτέρω συζητήσει. Έχουμε πληροφορίες για κάποια πειράματα που γίνονται στις περιφέρειες, ιδιαίτερες περιφέρειες που συμμετέχουν στο δίκτυο και μάλιστα είναι περιοχές με έντονη δραστηριότητα σε βιομηχανίες ε, τεχνολογίες διαστήματος. Αλλά οι εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης δεν ενδιαφέρουν μόνο αυτές τις περιφέρειες, αλλά όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Για παράδειγμα, το σχέδιο ή μάλλον το πείραμα που έγινε στη Βρέμη. για τον τρόπο διαχείρισης ε, μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια και τα θέματα ασφάλειας, ελέγχου διαχείρισης, είναι ένα πείραμα που είναι πολύ ενδιαφέρον από την άποψη εφαρμογών. Επίσης, ένα άλλο σχέδιο που αναπτύχθηκε για την πλοήγηση μεγάλης ακρίβειας σε λιμάνι είναι ένα πρόγραμμα που αποκαλείται Seagate, που χρησιμοποιείται στο Βόρειο Μπέγκελμπουργκ, η τελευταία περιοχή που προσχώρησε στον Ερέους, με το λιμάνι του Ροστόκ και αφορά τις εφαρμογές, ε, πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές για την ε, πλοήγηση μεγάλης ακρίβειας στα λιμάνια. Επίσης, ε, στη Βενέση έχουμε το πρόγραμμα Εξάντας, σε, σε που ελέγχει τις ροές κυκλοφορίας στις περιοχές ε, υψηλού κινδύνου κυκλοφορίας ή αιχμής κυκλοφορίας. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στις χερσαίες μεταφορές, αλλά και στις μεταφορές στις, στους αερολιμένες. Υπάρχει το σύστημα Κλέστα, για παράδειγμα, που αναπτύχθηκε στην Τουλούζη και στο στη ζώνη αερολιμένα του Μπορντό, που χρησιμοποιεί εφαρμογές για τη διαχείριση της ενέρειας κυκλοφορίας, αλλά και των υπηρεσιών ε, τεχνικής συντήρησης. Και υπάρχουν και άλλα σχέδια για τη βοήθεια ανθρώπων με προβλήματα κινητικότητας, για τη διαχείριση των ε, θέσεων στάθμευσης, για τα προβλήματα των τυφλών και στη Μαζοβία έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια στον τομέα της υγείας. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Θα ήθελα όμως να ολοκληρώσω με ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση. Πολύ συχνά οι περιφέρειες ε, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Και βρισκόμαστε στο στάδιο αυτό που θα αποκαλούσα ε, βιομηχανικό πειραματικό πρόγραμμα. Βέβαια, το θέμα είναι να περάσουμε από το βιομηχανικό πειραματικό πρόγραμμα στην εφαρμογή του στην αγορά και το πέρασμα από τον βιομηχανικό αυτοπιλότο στην αγορά χρήζει σημαντικής ε, και ταψιλούς χρηματοδότησης και σήμερα το ερώτημα που μας θέτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να γίνει αυτή η μετάβαση από το πείραμα, το βιομηχανικό πείραμα στην αγορά είναι η πιο αγκύρη ερώτηση και το θέμα της χρηματοδότησης αυτής της μετάβασης δυστυχώς δεν έχει επιληθεί. Αυτά γιατί μου ζητήσετε να είμαι λακωνικό, θα επανέλθουμε σε ορισμένα σημεία κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Darf mich äh, sehr herzlich bedanken. Να σας ευχαριστήσω. Κατόπιν η κυρία Πατάκη έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. ladies and gentlemen. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Σιγητά, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κανονισμός της ΕΝΣΕΣ ε, εκδηλήθηκε το 2008 και μεταμόρφωσε τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης και φέτος θα γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών και καλωσορίζω το ότι η Επιτροπή σας εδώ πέρα συντάσσει μια τέτοια έκθεση για να ακουστεί και το Κοινοβούλιο. Σήμερα θα αναλύσω τα αποτελέσματα, το τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής στον τομέα αυτών και κατόπιν θα προσπαθήσω να αναφερθώ στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας η απόφαση για το Γαλιλαίο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του 2008 άνοιξε τον ε, δρόμο και μπορούμε να πούμε για μια νέα αρχή και μπορούμε να πούμε πως ε, είχαμε μια επιτυχή απόφαση. Οπότε θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόν έγινε λοιπόν μια νέα αρχή, είχαμε μια επιτάχυνση και μια πιο διαφανή διαμόρφωση του προγράμματος, επίσης έγινε πιο δυναμικό και λειτουργούν καλύτερα και οι διοικητικέ δομές. Η Κομισιόν έχει ένα νέο ρόλο ως διαχειριστής του προγράμματος, κάτι το οποίο οδήγησε και στο απαραίτητο πλαίσιο. Η πολιετής ε, συμφωνία αντιπροσωπείας με την ΕΣΑ ξεκαθάρισε τον ρόλο και τις ευθύνες της ΕΣΑ ως ε, υπεύθυνου για τις προμήθειες και ως βασικού αναδόχου. Έχουμε λοιπόν την Επιτροπή του Προγράμματος και το διοργανικό πάνελ για το Γαλιλαίο που συνεργάζεται στενά με Κοινοβουλίο, Συμβουλίο και Κομισιόν. Τώρα όσον αφορά το Κοινοβούλιο, εκεί θα προτείναμε να εξεταστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά την επιτήρηση. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το καθεστώς του στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας, ξεκινώντας από την διαδικασία της Λισαβόνας και από την άλλη η σύσταση είναι να ενισχυθεί ο ρόλος ε, της ε, επιτήρησης στην ε, GIP και εάν ε, αποδειχθεί ε, κάτι τέτοιο απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνει και το Κοινοβούλιο της Αρμόδιας Επιτροπές του. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάτε πως το Κοινοβούλιο μέσω του GIP έχει αναλάβει την ευθύνη συνολικά για το πρόγραμμα. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης, ε, της κοινοτικής χρηματοδότησης, δηλαδή μέσω του κανονισμού GNSS, ε, κατέσε δυνατή την ενσωμάτωση και του έγνους και ξεκίνησαν οι προμήθειες του προγράμματος. Υπάρχουν έξι πακέτα εργασίας που ε, ορίστηκαν και υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο Αξιολόγησης η όλη διαδικασία προμήθειας FOC και βεβαίως έχουν ήδη βρεθεί η ανάδοχοι για αυτά τα πακέτα και στο πρώτο εξάμεινο του 2010 θα γίνει και η υπογραφή των ε, συμβάσεων. Τώρα υπάρχει βεβαίως ε, κάποια καθυστέρηση στην διαδικασία των προμηθειών, αλλά αυτό δεν διακινδυνεύει το πρόγραμμα το ίδιο. Εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να δούμε πως υπάρχει ισορροπημένη συμμετοχή της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12α του σχετικού κανονισμού. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία της διπλής προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 10α3D, 3Δ. Και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις όπως επίσης και στην διαδικασία του πακέτου 4 οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω το Κοινοβούλιο να δει πιο στενά αυτά τα ζητήματα. Τώρα όσον αφορά την διαχείριση του προπολογισμού να σας υπενθυμίσω πως με βάση την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να προετοιμάσει νέα επικαιροποιημένα νούμερα τα οποία λογικά θα συμπεριληφθούν σε αυτή την ενδιάμεση αξιολόγηση. Βεβαίως μπορούμε να έχουμε κάποιες ανησυχίες, για, κάποιες με για το μικρό περιθώριο που υπάρχει στην φάση FOC, κάτι το οποίο βεβαίω προκύπτει από το ότι η φάση IOV ξεπέρασε το προβλεπόμενο κόστος. Και θα θέλαμε και περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η κοινοτική χρηματοδότηση των 3.305 εκατομμυρίων ευρώ που συμπεριλαμβάνεται στα 400 εκατομμύρια που δόθηκαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Καλό θα ήταν να δει το κοινοβούλιο τι θα γίνει με αυτό το ποσό γιατί υπάρχει απολύτω απαραίτητη έρευνα που θα μπορούσε να επηρεαστεί όσον αφορά τώρα την πρόοδο στα συγκεκριμένα έργα είναι δύσκολο να κρίνουμε υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις όμως αυτό δεν βλάπτει την υλοποίηση των έργων δυστυχώς τα έγγραφα της Κομισιόν δεν συγκρίνουν το καθεστώς των έργων με το αρχικό σχέδιο εργασίας, οπότε δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το πώς πηγαίνουν τα έργα. Οπότε θα ήθελα να προτείνω να ζητήσει το Κοινοβούλιο πληροφορίες από την Κομισιόν. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν ήδη από τώρα όσον αφορά το έγνος. Μπορούμε να πούμε πως η διαδικασία της πιστοποίησης για την πολιτική αεροπορία ξεκινάει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο αυτό κανένα κράτος μέλος να μην βρεθεί στην θέση στην οποία δεν θα έχει πλήρη κάλυψη του σήματος σε ολόκληρη την επικράτειά του. Κάτι άλλο το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του GNSS θα πρέπει να περιέχει τα πρακτικά βήματα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να κατακτήσει την σχετική αγορά η οποία θα έχει αρκετά υψηλή αξία. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, στο δεύτερο μέρος ε, της συνεισφοράς μου θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα όσον αφορά τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε και εδώ πέρα να μένουμε τις ε, προτάσεις ε, της ε, Κομισιόν στο πλαίσιο της επερχόμενης ενδιάμεσης αξιολόγησης. Από όταν ξαναξεκίνησε το πρόγραμμα, το παγκόσμιο περιβάλλον έχει αλλάξει, η οικονομία έχει αλλάξει και η τεχνολογία έχει αλλάξει. Οι ανταγωνιστές μας, οι οποίοι βεβαίω είναι εν μέρη και εταίροι, αλλά κατά βάση είναι ανταγωνιστές, έχουν ενισχυθεί και υποθέτω πως σημειώνουν δυναμικές πρόοδους. Εδώ πέρα βεβαίως εγώ μιλάω για τα σχέδια εκείνα ναυτιλίας τα οποία προέρχονται από τον στρατιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει πως η παγκόσμια αγορά για το Γαλιλαίο περιορίζεται και η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση θα πρέπει να συγκεντρωθεί στα βασικά αυτά σημεία και να βρεθεί η κατάλληλη απάντηση όσον αφορά τώρα την διασφάλιση της χρήσης του Γαλλίου από την αγορά θα ήθελα να αναφέρω τα εξής. Πρώτον, το έγνος και το Γαλιλαίο είναι και τα δύο πολιτικά προγράμματα και οι, οι ανταγωνιστές μας έχουν στρατιωτικούς προϋπολογισμούς. Οπότε νομίζω καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε το PRS κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα βοηθούσε τα προγράμματα δορυφορικής ε, πλοήγησης. Επίσης η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από στήματα δορυφορικής ε, πλοήγησης σε πιο στρατηγικά παιδεία, κάτι το οποίο σημαίνει πως το σχέδιο δράσης θα πρέπει να επιταχυνθεί, παραδείγματο χάρη η τυποποίηση, η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει και αυτό την ε, δουλειά που του αναλογεί εδώ πέρα. Αυτό ούτως ή άλλως νομίζω αναφέρεται και στο 6α2 το άρθρο του σχετικού κανονισμού κατόπιν και τρίτον θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας εξαγωγικής πολιτικής στο Γαλιλαίο για να μπορέσουμε να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου στα ευαίσθητα ζητήματα. Τώρα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά καθήκοντα τα οποία προκύπτουν για τον ιδιοκτήτη του συστήματος. Ο ρόλος του ιδιοκτήτη του συστήματος είναι καινούριος για την κοινότητα, οπότε θα πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις. Μία απόφαση λοιπόν για την διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος μέχρι το 2013 είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά έχοντας υπόψη την προετοιμασία των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ε, πλοήγησης πλέον δεν αντέχουν καμία άλλη καθυστέρηση. Αλλιώς οδηγούμαστε σε τέλειο αντιέξοδο. Αυτό ίσχυε ήδη και το 2008 όταν απαιτήθηκε μία διόρθωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν γρήγορα να δούμε ποιες είναι οι εμπορικές πτυχές και οι νομικές συμβατικές πτυχές και η πτυχή της χρηματοδότησης. Κατόπιν, το ποιος έχει ναστική ευθύνη για την δορυφορική πλοήγηση, ειδικά σε σχέση με το έγνος, πρέπει να το δούμε για να μειωθεί ε, αυτή, ε, αυτός ο κίνδυνος σε περιπτώσεις όπου οι εφαρμογές αυτές είναι κρίσιμες για την ασφάλεια. Και τέλος, ειδικά στοιχεία του συστήματος ε, λείπουν ακόμα, π.χ. ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαχείρισης του κινδύνου, σημεία απολύτως απαραίτητα που προκύπτουν για τον ιδιοκτήτη του συστήματος. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δορυφορικής πλοήγησης. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές πλοήγησης και τις υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως αυτό είναι κάτι ξεχωριστό από το πρόγραμμα GNSS, αλλά νομίζω πως ε, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σωστά χωρίς μια τέτοια συμφωνία. Και βεβαίως ως άμεσα εκλεγόμενο σώμα της ε, κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, τελείωσε ο χρόνος μου. Ελπίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτά τα προγράμματα. Είναι μια στρατηγική αποστολή και θα εξακολουθεί να παίζει τον ηγετικό του ρόλο στην διαδικασία. Και με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βάρση Πατάκη. Ο κύριος Τορτόρα έχει τώρα τον λόγο. Uh, <clears throat> so, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνθηκε να εκφράσω τις απόψεις του κλάδου για το σημαντικό αυτό πρόβλημα, ε, το Χαλιλαίο δηλαδή, στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή στην πορεία της ιστορίας του. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι το 2008 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε έναν έλεγχο, διεξήγαγε έναν έλεγχο και αξιολόγησε το, την ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο έλεγχος ήταν σημαντικός. Δεν θα επισέλθω στα απορίσματα και στις ε, συστάσεις που εκδόθηκαν τότε, αλλά θα υπογραμμίσω κατά πόσο η ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων, η διαχείριση των προγραμμάτων είναι ένα δύσκολο καθήκον και η ανοικοδόμηση ε, διαχειριστικών ικανοτήτων είναι κάτι που πρέπει να το ξεκινήσουμε από την αρχή και μας θέτει πάρα πολλές προκλήσεις. Έκτοτε έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και θα ήθελα να, από, ζητήσω φόρο τιμής κατά κάποιον τρόπο προς την Επιτροπή και το προσωπικό της για την διαχείριση των δραστηριοτήτων του Γαλιλαίου. Αλλά σήμερα φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει κυρίως το ενδιαφέρον της στον έλεγχο των κονδυλίων, στους ελέγχους και τις διαδικασίες, στα, στα νομικά και διοικητικά καθήκοντα εν ολίγης. Από την οπτική της βιομηχανίας του κλάδου μοιάζει σαν να υπάρχει έλλειψη ε, διαχειριστικής ικανότητας των προγραμμάτων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Η διαχείριση προγραμμάτων τι είναι. Ένα πρόγραμμα ε, πρέπει κανείς να το διαχειριστεί κατά κάποιον τρόπο, καταρχήν πολιτικά. Όλοι αναμένουμε ένα έντονο τέτοιο πολιτικό σήμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όμως να διαχειρίζεται και τεχνικά. Και ε, εδώ σίγουρα μπορούμε να παρέχουμε εμείς στήριξη στην Επιτροπή. Επίσης πρέπει να διαχειριστεί και από βιομηχανική άποψη. Και από αυτήν την άποψη ε, χρειάζεται μια προσαρμογή των κοινοτικών, των ενωσιακών κανόνων. Από πολιτική άποψη η ΕΣΑ μπορεί να παρέχει στήριξη, σίγουρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μπορεί να, δεν μπορεί να θεσπίσει τους στόχους του προγράμματος η ΕΣΑ, αλλά σίγουρα μπορεί πολλά πράγματα να κάνει. <clears throat> Ε, κοινότητα, η Ένωση έχει σίγουρα το βασικό ρόλο να παίξει στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά οι κανόνε και οι δομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταπακριθούν καλύτερα στις βιομηχανικές, στη, στην πραγματικότητα τη βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για δικηγόρους να συνεννοούνται με μηχανικούς. Όλοι το ξέρουμε αυτό και η διαχείριση ενός προγράμματος δεν είναι δυνατόν να τοποθετείται μόνο στο δημοσιονομικό ή στο χρηματικό ή στο οικονομικό επίπεδο. Πρέπει κανείς να ξέρει τον κλάδο, να γνωρίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο κλάδος. Και πίσω από κάθε απόφαση αυτό που διακυβεύεται είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων και δυναμικότητας στον διαστημικό χώρο. Αυτή η ικανότητα είναι κάτι που θα καθορίσει ε, την κυριαρχία της Ευρώπης και την αυτονομία της στον ε, χώρο και στο διάστημα. Η διαχείριση του προγράμματος ε, Γαλιλαίου καθεαυτή τώρα. Ε, γράφω εδώ δεξιότητες του προσωπικού, ενώ δεξιότητες του δημόσιου προσωπικού. Αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβει όλους τους τομείς. Θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικές ικανότητες, νομικές, διαχειριστικές, εμπορικές, επιστημονικές, οικονομικές, βιομηχανικές. Πώς θα καλυφθούν όλες αυτές οι δεξιότητες. Σίγουρα δεν είναι η βιομηχανία που θα υπαγορεύσει πώς πρέπει να οργανωθεί ο δημόσιος τομέας, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως ε, θα πρέπει ε, να βασιστούμε περισσότερο στην ΕΣΑ. Υπάρχουν και οι δύο επιλογές ε, ανοιχτές σήμερα. Το δεύτερο αφορά την σταθερότητα του προσωπικού γιατί η ικανότητα του προσωπικού, οι ικανότητες του προσωπικού είναι κάτι το οποίο χτίζεται με το χρόνο. Ε, σίγουρα απαιτείται κάποια σταθερότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί και να ενισχυθεί ε, η ικανότητα του, του προσωπικού του δημόσιου τομέα. Η το να υπάρχει ένας υψηλός ρυθμός εναλλαγής στα πόστα αυτά ε, υπονομεύει την σταθερότητα και, την, και μια πραγματική ικανότητα διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να εξατομικευτούν οι διαδικασίες ε, για μια αποτελεσματική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων η διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερότητε των διαστημικών προγραμμάτων και σίγουρα σε μερικούς μήνες από τώρα θα πρέπει να ξαναδούμε την όλη διαδικασία των ε, δημόσιων προμηθειών. Και τέλος θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη ανάθεση αρμοδιοτήτων και παραχώρηση αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους στη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Πέρα από το Γαλιλαίο, γιατί το πρόγραμμα Γαλιλαίος ασφαλώς θα διαμορφώσει το μέλλον και τις μελλοντικές ε, ικανότητες, τη μελλοντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χειριστεί όλα τα ε, διαστημικά ενδιαφέροντα και τις δομές που σχεδιάζονται. Υπάρχει το Caesar, ο Κέσαρας, για την ενέργεια κυκλοφορία, το GMES ε, για παρατήρηση. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν και θέματα για την επίγνωση της ασφάλειας στο διάστημα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει ασφάλεια κατά την εκτόξευση δορυφόρων στο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ικανότητα της εξασφάλισης της ορθής διαχείρισης όχι μόνο της φάσης εξέλιξης των προγραμμάτων αλλά και της επιχειρησιακής ε, δραστηριότητας των προγραμμάτων. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη ε, οι σχετικοί κανόνες θα έχουν ε, θα παίξουν μεγάλο ρόλο γιατί ανοίγεται έστω και μια περιορισμένη εμπορική αγορά. Θα περάσω στα συμπεράσματα. Ο κλάδος χρειάζεται ένα αρμόδιο, ένα ικανό δημόσιο σύστημα. Ο πελάτης ξέρει τι θέλει, ε, θέλει να το βρει και αυτό που θέλει ο κλάδος είναι να υπάρχει ένα και μόνο σημείο συνεννόησης με τους ε, δημόσιους ε, θεσμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε τώρα και τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Στάρεκ που πρέπει να αλλάξει, νομίζω θέση στον υπολογιστή. Ε. Περιμένουμε ένα λεπτάκι. So, good afternoon. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε μέλη, βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να πάρω μέρος σε αυτή την ακρόαση, γιατί, ο τομέ... γιατί μας ενδιαφέρουν όλες οι δραστηριότητες και οι δράσεις που εντάσσονται στην προβληματική των ευρωπαϊκών συστημάτων πλοήγησης και, και σχετικών τεχνολογιών ε, μια σύντομη εισαγωγή, να συστηθώ. Είμαι ο Τόμας Στάρεκ, ε, εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο στην Πράγα και εργάζομαι και στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η παρουσίασή μου λοιπόν θα εστιαστεί περισσότερο στην χρήση των σχετικών εφαρμογών και την σημασία της χρήσης του Γαλιλαίου και την ε, εφαρμογή του. Εδώ βλέπετε κάποιους τομείς ε, που ωφελούνται από το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Έχοντας αυτό κατά νου, ε, θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες δραστηριότητες που βρίσκονται στο προεπιχειρησιακό στάδιο, καθότι η εξέλιξη και η σχεδίωση του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί. Στη φάση αυτή πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά την πιθανή, την πιθανή ανάμειξη επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Γαλιλαίου. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες βιώσιμες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ρόλο, θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να, γίνουν να υπάρχουν εφαρμογές στα διάφορα επίπεδα των υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από το Γαλιλαίος. Αυτό τι σημαίνει. Σε ένα επίπεδο, στο επίπεδο 1, έχουμε την ανοιχτή λειτουργία του Γαλιλαίου, η οποία πέφτει σε, ε, η οποία στην κατηγορία των εφαρμογών που δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Ε, μετά υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες εναέρειας κυκλοφορίας και αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για την πιθανή ανάμειξη και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στα διάφορα επίπεδα των υπηρεσιών του Γαλιλαίου. Ε, υπάρχουν ε, διάφοροι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για, να, για να υποφεληθούν οι χρήστες από τις εφαρμογές του Γαλιλαίου. Αφού έχουμε κάνει αυτή τη χαρτογράφηση μεταξύ των εφαρμογών των υπηρεσιών του Γαλιλαίου, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας έντονα σε μια ανάλυση της αγοράς από την άποψη των εφαρμογών, που θα καλύψουν όχι μόνο τη σημερινή κατάσταση, αλλά και τις προοπτικές. 50 συν, ε, μετά το 2015. Εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια το 2009 από το GNSS, ε, εφαρμόστηκε ε, το παρατηρητήριο αγοράς GNSS, το οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την πρόβλεψη συμπεριφοράς της αγοράς GNSS στην Ευρώπη. Και πάνω σε αυτή τη βάση θα μπορέσουμε πιστεύω να προετοιμαστούμε καλύτερα για διάφορα επιχειρηματικά σενάρια. Αυτό το λογισμικό βασίζεται σε διάφορες πηγές δεδομένων και διάφορες παραδοχές. Ε, βασικά προέρχονται από το, από μελέτες ε, του GSA, από προγράμματα πλαίσιο ε, για την έρευνα και την τεχνολογία. Εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να ορίσουμε τους διάφορους όρους χρήσης για τα διάφορα επίπεδα υπηρεσιών του Γαλιλαίος και πρέπει να κάνουμε μια αρχική ερώτηση. Τι πραγματικά αναμένουμε, τι, ποια θεωρούμε ότι είναι κάποια βιώσιμα επιχειρηματικά σενάρια, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Μπορεί να πει κανείς είτε ναι, θέλουμε να έχουμε βιώσιμα επιχειρηματικά σενάρια για το επιχειρησιακό στάδιο εφαρμογής του Γαλιλαίος, ε, ή μπορούμε να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε τέτοια σενάρια και αυτό έχει μεγάλη διαφορά για το πώς θα διαχειριστούμε τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη γιατί και οι δύο εφαρμογές για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ο Γαλιλαίος στο μέλλον ε, θα, θα είναι ανοιχτέ στο κοινό, θα χρησιμοποιηθούν από το κοινό. Επομένως θα είναι ένα δημόσιο όφελος και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες του, αυτού του δημόσιου ωφέλους. Μπορούμε να πούμε ε, είτε ότι δεν χρειαζόμαστε τέτοια βιώσιμα ανεξάρτητα επιχειρηματικά ε, σενάρια ε, ή αν θα αποφασίσουμε να καλύψουμε αυτά τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη για να καλύψουμε μάλλον τα κοινωνικονομικά ωφέλη ή εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θα διαχειριστεί αυτά τα ωφέλη. Ανέφερα νωρίτερα την μελέτη GNSS και την αγορά GNSS, ε, ε, όπου ένα μεγάλο μέρος των του σχετικού κοινωνικο-οικονομικού ωφέλους ε, το απολαμβάνει ο τομέας των σιδηρόδρομων. Αλλά θα μπορούσαμε να εντάξουμε και άλλους τομείς, τη γεωργία, ε, τη αέρια κυκλοφορία, ε, τις τηλεπικοινωνίες. Βλέπετε ότι διακυβεύονται πολύ μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το χειριστούμε στα διάφορα επιχειρηματικά μας σενάρια. Όσο αφορά τις ευκαιρίες αγοράς ε, κατά την περίοδο από τώρα μέχρι το 2015, μπορεί κανείς να αναμένει μια αύξηση εφαρμογών που θα καθοδηγούνται κυρίως από το κανονιστικό πλαίσιο. Έχουμε την, ε, τις διάφορες οδηγίες για τα, τις ηλεκτρονικές οδηγίες, επίσης την ε, οδηγία για τις μεταφορές, η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Έτσι μπορεί να δοθεί μια όθηση στη χρήση του προγράμματος Γαλιλαίος και να δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση χρηστών. Και ακόμα πιο σημαντικό θα υπάρχει δυνατότητα για υπηρεσίες πρόσθετης αξίας, οι οποίες στη συνέχεια θα καλυφθούν από τις ανοιχτές υπηρεσίες του Γαλιλαίου. Τώρα, αυτές οι εφαρμογές οι οποίε θα καθοδηγούνται κατά κάποιο τρόπο το κανονιστικό πλαίσιο, λόγω ε, <clears throat> της έντονης ε, τοπικότητας των εφαρμογών, υπάρχουν κάποια συστήματα αυτή τη στιγμή που υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να αναφέρω το Civis Κούπερς και άλλους, οι οποίοι ασχολούνται με ένα σύστημα συνεργασίας και ένα σύστημα αυτόματης παροχής σύνδρομης στον τομέα των ε, αυτοκινητιστικό. Εκεί ε, πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί μια μεγάλη πελατειακή βάση για το Γαλιλαίος. Και τέλος, αλλά όχι γενικότερο σημαντικό, υπάρχουν ειδικέ εφαρμογές. Αστρατιωτικές εφαρμογές, οι οποίες αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και εντατικά. Επίσης, ε, διάφορες εφαρμογές ενοποιημένης αντιμετώπισης κινδύνων, έλεγχος των αεροπορικών ε, έλεγχος των αεροδρομίων, των διαδρόμων τροχοδρόμησης, πλοήγηση σωστικών ε, σωμάτων, σωμάτων διάσωσης, Υπάρχει μια έμφαση σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσει συστήματος στις ρυθμισμένες υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα εξυπηρετηθούν από το Γαλιλαίος. Η ιστορία με τις ευκαιρίες της ΑΓΟ υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία για τις ευκαιρίες αγοράς. Είναι μια τεράστια εμπορική αγορά, ιδίως στην ε, πλοήγηση των αυτοκινήτων, στην, ε, στα προϊόντα Pay As You Drive, διάφορα προϊόντα που βρίσκονται εν εξελίξει στην Ευρώπη. Ε, ξέρετε πόσο έντονη είναι η θέση του GPS στην αγορά και είναι δύσκολο να πιστούν οι χρήστες να αγοράσουν καινούριο εξοπλισμό τώρα ή να περάσουν σε καινούρια συστήματα, να έχουν και πομπούς ε, γαλιλαίος. Εγώ όπως το βλέπω είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, ιδίως για το marketing, πώς θα παρουσιαστούν τα ωφέλη του γαλιλαίου στην πράξη. Αυτό μπορεί να είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να αρχίσουμε αμέσως με θετικές εκστρατείες ε, που θα παρουσιάζουν στους χρήστες των υπηρεσιών του Γαλιλαίος ε, το περιεχόμενο και τα διάφορα ωφέλη που θα έχει. Θα ολοκληρώσω τώρα την παρουσίασή μου. Προετοίμασα την τελευταία διαφάνεια, η οποία είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες. Θέλω να τονίσω εδώ ε, από τη θέση αυτή ότι ε, το πρόγραμμα Γαλιλαίος αναφέρεται πάντοτε ως ένα πολύ ωφέλιμο τμήμα των υπηρεσιών, ότι προσφέρει υψηλή αξία στις παραμέτρους του συστήματος. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως ανέφερα στην πλοήγηση αυτοκινήτων, είναι αλήθεια ότι πραγματικά συνεισφέρει πολύ ο Γαλιλαίος, το πρόγραμμα Γαλιλαίος σε αυτές τις εφαρμογές και οι παράμετροι του συστήματος ε, του προγράμματος Γαλιλαίος θα, θα επηρεάσουν έντονα τις επιδόσεις ε, των εφαρμογών. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και ένα είδος ε, μιας άλλης ασύρματης επικοινωνίας. Εδώ έχω βάλει επικοινωνία μεταξύ δύο αυτοκινήτων. Επικοινωνία μεταξύ δύο αυτοκινήτων. Και αν δούμε αυτήν την εικόνα θα, θα καταλάβουμε ότι για να εκπληρωθούν όλες οι εφαρμογές και οι παράμετροι των συστημάτων το ζήτημα δεν είναι μόνο η επικαιροποίηση τοπικά των διαφόρων ε, παραμέτρων αλλά έχουμε και το, τη διάσταση των τηλεπικοινωνιών, γιατί είναι, και έχει ζωτική σημασία αυτό, γιατί μπορεί να έχεις μια ωραία εφαρμογή στο τέλος που να φαίνεται τέλεια και, και σούπερ, αλλά και μπορεί όμως να έχεις δείκτες επιδόσεων ε, όσο αφορά τη χρήση που να είναι πολύ κακές, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη ε, οι διαστάσεις των τηλεπικοινωνιών. Τώρα, εν κατακλείδη, έχω συνοψίσει εδώ κάποια βήματα τα οποία μπορεί να μας οδηγήσουν σε, μια καλή, σε ένα καλό επιχειρηματικό σενάριο Νομίζω ότι είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν ε, ουσιαστικά σε αυτήν την ε, φάση προετοιμασίας των επιχειρήσεων, να δώσουν στοιχεία, να, να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του παρατηρητηρίου της αγοράς GNSS, να κατατάξουν τις διάφορες εφαρμογές σε κατηγορίες, να υπάρχει έντονη επικέντρωση στα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την δορυφορική πλοήγηση και τις σχετικές τεχνολογίες, γιατί αυτά δείχνουν ποια θα είναι η μελλοντική χρήση του Γαλιλαίος. Και τέλος, όπως είπα και στην προηγούμενη διαφάνειά μου, καλό είναι να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας την τελική, τις τελικές επιδόσεις του προγράμματος ε, και την ανάγκη κάλυψης και των άλλων διαστάσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις ε, εμπειρογνώμονες και γιατί τηρήσατε το χρόνο. Οπότε έχουν τώρα οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να κάνουν ε, ερωτήσεις. Ε, έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ρωτήσετε τους ειδικούς μας. Κύριος Μποριζίνα πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που υπάρχει κάποια πρόοδος επιτέλους και βλέπουμε να γίνονται επιτέλους τα πρώτα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην εφαρμογή του προγράμματος Γαλιλαίου. Βέβαια είναι πολύ φιλόδοξο και απαιτητικό αυτό το πρόγραμμα και έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τις εφαρμογές αλλά και για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν πολλά ωφέλη από το σύστημα αυτό. Δεν είναι μόνο οι εφαρμογές του, αλλά και οι τεχνολογίες που θα εφαρμόσουμε. Και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Είναι πολύ χρήσιμε ε, οι πληροφορίες που ακούσαμε για το πρόγραμμα Νερέους και περιμένουμε και γραπτός τεκμηρίωση. Μου άρεσε πολύ και η παρουσίαση της κυρίας Μπάρση Πατάκη την γνωρίζουμε άλλωστε από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, την κυρία Πατάκη. Και το όνομά της ουσιαστικά συνδέθηκε άρρηκτα με το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Για να μην σας πω ότι όταν ακούμε Γαλιλαίο μας έρχεται ως εξίσωση αμέσως και το όνομα της κυρίας Μπάρση Πατάκη. Σε ό,τι αφορά την ε, παρουσίαση του κυρίου Τορτόρα, όταν διάβασα τη μελέτη για το πρόγραμμα Γαλιλαίος, δημιούργησε την εντύπωση ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είχε σαφή διαχειριστική δομή ακόμη σε όλα τα επίπεδα. Και δυστυχώς ε, η παρουσία του κυρίου Τορτόρα δικαίωσε αυτή την εντύπωση που σχημάτισα. Φαίνεται ότι είναι απροσδιόρισες ακόμη οι διαχειριστικές δομές του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές που παρουσιάστηκαν, από τους εμπειρογνώμονες και οι δυνατότητες ε, χρήσης των τεχνολογιών αυτών που μέχρι στιγμής δεν αξιοποιήθηκαν δυστυχώς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εμπειρογνωμονές μας για τις πληροφορίες αυτές, γιατί είμαι ο σκιώδης ηγητής του κόμματο μου για το θέμα αυτό και θα ήθελα εκ βάθους καρδίας να σας ευχαριστήσω θερμά για την πλούσια ενημέρωση. Το ερώτημά μου αφορά την ε, οργανωτική δομή του προγράμματος. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα χάρη σε καλύτερη οργανωτική δομή. Υπάρχουν αποκρισταλωμένες απόψεις για την οργανωτική δομή που απαιτείται για την προώθηση αυτού του προγράμματος. Βέβαια, παρά είναι ευρύ το πεδίο αυτού του ερωτήματος, ίσως μπορείτε να με παραπέμψετε σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία για να ενημερωθώ. Γιατί γνωρίζω ότι τέτοια πολυσύνθετα προγράμματα πρέπει να στηρίζονται σε στερεή οργανωτική βάση. Και αυτό το πρόγραμμα είναι από τα πιο περίπλοκα που είδαμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερα μια τέτοια βάση. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ειδικού μας. Με συγχωρείτε για το ότι άργησα και άκουσα μόνο τον... την τελευταία παρέμβαση αλλά ήταν και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα εγώ από την πολιτική πτυχή να σας ρωτήσω ποια είναι τα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να θέσουμε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Απευθύνομαι εδώ πέρα στον τελευταίο μιλητή που μιλάει για τα προπαρασκευαστικά μήματα της επιχειρησιακής φάσης. Θέλουμε ένα σύστημα Γαλιλαίο το οποίο θα είναι αποδοτικό με οικονομικές ε, υπηρεσίες ή μήπως μακροπρόθεσμα ή και πάντα θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί μόνο με την υποστήριξη του φορολογουμένου. Είναι αυτό το βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε ως πολιτική πέραν των άλλων ερωτημάτων που έθεσε η κύριε συνάλφος, δηλαδή τι θα κάνουμε με τα ζητήματα διαχείρισης, αλλά... Το ερώτημα για μένα είναι πώς θα μπορούσε να είναι οικονομικά αποδοτικό και να στηρίζεται στα δικά του τα πόδια το Γαλιλαίο τελικά. Ε, το θεωρείτε κάτι τέτοιο ρεαλιστικό, αν θυμηθώ και την προϊστορία του Γαλιλαίου, το οποίο το είχαμε δει στο πλαίσιο μιας ΣΔΙΤ ε, πριν από 10 χρόνια ακόμα. Θυμάμαι πως έλεγαν πως δεν υπήρχε επιχειρηματικό σχέδιο που θα λειτουργήσει εξού και καταλήξαμε στη ΣΔΙΤ, η οποία όμως επίσης δεν επέτυχε και καταλήξαμε τελικά στη δημόσια χρηματοδότηση. Οπότε, υπάρχει κάποιο σενάριο ε, στο οποίο τελικά θα έχει κάποιες εισπράξεις ε, ο Γαλλίος και θα πατάει στα πόδια του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Έντσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. οι εμπειρογνώμονές μας πότε πιστεύετε ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Και η δεύτερη ερώτηση που εμπεριέχει και μια πρόταση. Τι χρειάζεται για να γίνει βιώσιμο και οικονομικά το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς που είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, θα μπορούσαν να επιβάλλουν στους κατασκευαστές συστημάτων μεταφορών να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Γαλιλαίο για να δικαιολογήσουμε τις τεράστιες επενδύσεις που κάναμε στο πρόγραμμα αυτό και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την ε, αυτάρκεια του την οικονομική, τη χρηματοδοτική. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να ξαναδώσω τον λόγο στου τέσσερι ειδικού, ξεκινώντα από την κυρία Πατάκη. Ε, ε, Επιτρέψατε μου να απαντήσω αμέσως στα ερωτήματα των συναδέλφων Μπρεζίνα και Νίμπλερ. Όπως είπα στην ε, παρουσίασή μου, η οικονομική και τεχνολογική κατάσταση παγκοσμίω έχει αλλάξει από όταν ξεκινήσαμε τον Γαλιλαίο. Κατά την άποψή μου πρέπει, πρέπει αυτό να το δεχτούμε, να το λάβουμε υπόψη. Οι ανταγωνιστές μας έχουν όλοι στρατιωτικούς προϋπολογισμούς. Έχουν τη δυνατότητα, έχουν ε, μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης. Αυτό το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα είναι το PRS να στηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα γιατί αυτό θα μπορούσε να συγκρατήσει, να στηρίξει το σύστημά μας. Είναι βεβαίως ένα πολιτικό σύστημα, μη στρατιωτικό, αλλά παρόλα αυτά συγχρηματοδοτείται ή θα έπρεπε να συγχρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό νομίζω πως είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Από την άλλη, έχουμε ένα έγγραφο της ε, Κομισιόν, ε, το οποίο φορά το σχέδιο, το πρόγραμμα εργασίας 2010 και εκεί πέρα αναφέρεται πως πρέπει πολιτικά να αποφασίσουμε τι μοντέλο θέλουμε για την επιχειρησιακή φάση. Και μετά η Κομισιόν θα μας προτείνει τα ζητήματα της αστικής ευθύνης, τα διάφορα ανοιχτά ζητήματα. Νομίζω πως εμείς ήδη από πλευράς Κοινοβουλίου πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα τι δυνατότητες έχουμε, τι ευθύνη θα πρέπει να αναλάβουμε στον τομέα της αστικής ευθύνης και μετά μπορούμε να αποφασίσουμε τι μοντέλο θέλουμε. Για εμένα ένα δεύτερο ερώτημα είναι εάν έχουμε και αν θα έχουμε αρκετά έσοδα μέσω του Γαλλίου. Για μένα το μεγαλύτερο ερώτημα πάντα είναι τι ευθύνη θα έχουμε και εμείς θα υπομισθούμε ως δημόσιους τομέας. Κατά την άποψή μου και αυτό ίσως απαντάει την ερώτηση το τι δομή πρέπει να έχουμε όπως το έχω δει εγώ πιθανώς ε, στην ε, επιχειρησιακή ε, φάση να επιλέξουμε ένα δημόσιο μοντέλο. Νομίζω πως όλες οι νέες τεχνολογίες πρέπει να λειτουργήσουν για αρκετά χρόνια μέχρι να αποδειχτεί 100% πως λειτουργούν και τότε ίσως να συμπεριλάβουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι απολύτως απαραίτητο για την πρώτη επιχειρησιακή φάση για αρκετά χρόνια να στηριζόμαστε και να μείνει αυτό το έργο στο δημόσιο τομέα. Βεβαίως το θέμα είναι τι κοστίζει. Και νομίζω πως εδώ πέρα η Κομισιόν πρέπει να μας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Και μετά μπορούμε να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπενετό. Θα επανέλθω και εγώ στο θέμα της χρηματοδότησης, γιατί το δίκτυο Νερέως ε, ασχολείται με όλα τα προγράμματα εφαρμογής ε, τεχνολογιών διαστήματος. Το GNSS είναι ένα από αυτά. Και πριν δύο-τρία χρόνια προβληματιστήκαμε για τη χρηματοδότηση του GMS. Και μάλιστα τότε υπό Αυστριακής Προεδρίας ασκήθηκε μεγάλη πίεση να αντιληφθεί η χρηματοδότηση του GMS e από ιδιωτικά κονδύλια. Βέβαια αυτό είναι πιο προφανές στο GMS e από ό,τι στο Γαλιλαίο και στο GNSS. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι αν περιμέναμε ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη τέτοιων αποστολών που θα είναι κοινοφελείς, θα έχουν κοινοφελή χαρακτήρα κρατικό, το θέμα τη πρόληψη των κινδύνων και όλα αυτά, γιατί για το GMS υπήρχε αυτό έντονα, αλλά για τον Γαλιλαίο με εντυπωσιάζει η σημερινή συζήτηση. Γιατί το θέμα για τον Γαλιλαίο δεν τέθεται με τους, ίδιου όρου, ίδιους όρους από ότι για το GMS. Και μάλιστα τότε ο Επίτροπος Βερχόγγεν σε μια συνεδρία στη Λιλή είχε εξαγγείλει το 2012-2013 την ε, δωρεάν χρήση των δορυφορικών δεδομένων και την ε, ανάπτυξη των εφαρμογών. Και σήμερα υπάρχει το πρόγραμμα DORIS στα πλαίσια του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, όπου 7 ή 8 περιφέρειες που είναι και μέλη του Νερέους, με επικεφαλής της αιών της Βρέμης, ε, εφαρμόζουν κάποια πιλωτικά προγράμματα για να δουν πώς θα προετοιμαστούν για το 2012-2013 όταν θα εξασφαλιστούν τα κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τη χρήση των δεδομένων. Τώρα βέβαια είμαστε ακόμη στο 2010 και το πρόγραμμα Doris αναζητεί κρατικά κονδύλια ή περιφερειακά ή κρατικά ή κοινοτικά από τα διαρθρωτικά ταμεία για να, γίνουν, για να αναπτυχθούν εφαρμογές του GMS και η συζήτηση για το Γαλιλαίο ίσως ε, τίθεται με άλλους όρους, γιατί εκεί όταν μιλούμε για μεταφορές ή για ε, εφαρμογές στη γεωργία ή για θαλάσσιες μεταφορές, ναυτιλία, πολύ πιο εύκολα, και αυτό δείχνει και η συζήτηση ε, ότι δεν είναι σωστό, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε επιχειρηματικά συμφέροντα στο Γαλιλαίο από ότι στο JMS φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται η συζήτηση για το Γαλιλαίο όπω είχαμε και για το GMES. Ελπίζω το συμπέρασμα να είναι το ίδιο, ότι θα πρέπει να περάσουμε από κρατική χρηματοδότηση, δημόσια χρηματοδότηση, αν θέλουμε να αναπτύξουμε τι εφαρμογές. Δεν ξέρω κυρία Μπάρση Πατάκη πότε θα καταλήξουμε σε αρμονική και θετική ανάπτυξη για να προσελκύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια σε εφαρμογές που θα έχουν ε, δείξει ότι είναι χρήσιμες και σωστές έχω ένα ερωτηματικό για αυτή την θεωρία. Πάντως το θέμα της χρηματοδότησης ε, που θα είναι η κρατική ή η δημόσια, η δημόσια ή η δημοσια η είναι στο επίκεντρο της ε, συζήτησης. Πότε θα είναι επιχειρησιακό το και λειτουργικό το πρόγραμμα. Πριν από λίγο σας ανέφερα ε, μία παρατήρηση ομάδα εργασία για το GNSS του Νερέους. Χρειαζόμαστε χένκια και για το θέμα τη διακυβέρνηση. Πώ θα λειτουργήσει το σύστημα, Αυτό προβληματίζει και τις περιφέρειες, αλλά και τους ε, επιχειρηματίες και τους τοπικούς παράγοντες. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και πώς όλα αυτά τα προγράμματα θα εφαρμοστούν και ποιος θα τα κατευθύνει, ποιος θα τα χειριστεί. Σίγουρα θα πρέπει προηγουμένως να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα και για το Γαλιλαίο. Πότε θα είναι δηλαδή λειτουργικό επιχειρησιακό το Γαλιλαίο. Ευχαριστώ κύριο Στορτόρα. Ευχαριστώ. Εστερνίζομαι τις απόψεις των προλαλισσάντων σε ό,τι αφορά τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού κλάδου για το θέμα του Γαλιλαίου. Και μάλιστα αυτή ήταν και από τις γενισουργές ε, ιδέες του προγράμματος Γαλιλαίο και έδειξε τα όρια της και μας έφερε σε διέξοδο όταν προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για την ανάπτυξή του. Και Χαίρομαι για τις θεραλές απο, αποφάσεις που ελήθησαν για να επανέλθουμε σε 100% θεσμική κρατική δημόσια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε επιτέλους ε, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα Γαλλία. γιατί αν περιμέναμε από τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν επρόκειτο να γίνει. Σε ό,τι αφορά το GMES, η ίδια συζήτηση είχε γίνει και τότε και είναι αναφίβολο σήμερα, αναφισβήτητο, ότι το μέσο και και μέσο πρόθεσμο μέλλον του Γαλιλαίος ε, στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση, στη δημόσια χρηματοδότηση και όχι στην ιδιωτική. Τώρα, πότε θα είναι επιχειρησιακό το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Θα ήθελα να δείξω μια αισιοδοξία σήμερα, γιατί πιστεύω ότι η πιο δύσκολη φάση ήδη πέρασε. Γιατί το πιο δύσκολο ήταν να ληφθεί η απόφαση. Η απόφαση ελήφθη και τώρα απομένει το πιο δύσκολο τεχνικό, βιομηχανικό και τεχνολογικό σκέλος. Αλλά εδώ είμαστε σε σφαίρες και δραστηριότητες πολύ πιο γνωστές που επιδέχονται προγραμματισμού, σχεδιασμού. Οπότε μπορούμε να επιδείξουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία και να έχουμε εμπιστοσύνη στις προθεσμίες υλοποίηση αυτής της φάσης. Αλλά αυτά για την υποδομή της θέσης τροχιά. Πέραν τούτου όμως θα πρέπει να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες για να γίνει πλήρως ε, λειτουργικό το σύστημα, το δορυφορικό και να φτάνει και μέχρι τον τελικό χρήστη. Πάντως ε, είναι τεράστιο το έργο που έχουν να, να κάνουν τώρα οι βιομηχανίε για το θέμα αυτό. Ο κύριο Στάρεκ. Takže, a pánové, já nejprve rád odpověděl na otázku související s financováním a... Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, να πω δύο λόγια για τη χρηματοδότηση. Σίγουρα μιλούμε κυρίως για δημόσια χρηματοδότηση, γιατί το επενδυτικό και αναπτυξιακό τμήμα του Γαλιλαίου χρηματοδοτείται από δημόσια κονδύλια, γιατί το πρόγραμμα PPP απέτυχε στον τομέα αυτό. Το, το θέμα της σύμπραξης δηλαδή ιδιωτικών και δημόσιων κονδύλιων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή φάση, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές παράμετροι για τις υπηρεσίες του Γαλιλαίου. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βρούμε το κατά πόσο θα είναι οικονομικά βιώσιμο αυτό το πρόγραμμα, αν μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί ή τι άλλα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη μπορεί να επιφέρει. Ελπίζουμε να ανθίσει η αγορά για το GNSS. Αλλά όλα τα στοιχεία που έχουμε ακόμη είναι πολύ γενικά. Και σίγουρα δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε ένα καταμερισμό των ωφελών μεταξύ των διαφόρων ε, υπηρεσιών ή τομέων που θα καλύψει το σχέδιο Γαλιλαίο. αν η δημόσια χρηματοδότηση του Γαλλίου στηριχθεί σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, θα είναι καλό, αλλά και κάποιες κοινοφελείς υπηρεσίες. Βέβαια θα πρέπει να δούμε τι μερίδιο της αγοράς καλύπτει. Τι μερίδιο της αγοράς καλύπτουν αυτές οι υπηρεσίες, οι κοινοφελείς, σε σχέση με τις ανοιχτές ή εμπορικές υπηρεσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι για να έχουμε μία σαφέστερη εικόνα για τα οικονομικά ωφέλη του Γαλιλαίου, θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε ένα καταμερισμό μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, το διαχειριστικό σκέλος του Γαλιλαίου, που ήταν και η πρώτη ερώτηση που τέθηκε, Όντως είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα και η διαχείριση του προγράμματος αυτού προαπαιτεί ένα συντονισμό σε πολλά επίπεδα. Αυτά μας ανέπτυξε ο Στορ τώρα στην ε, παρουσίασή του. Και πιστεύω ότι η λειτουργία του GSA είναι ένα καλό παράδειγμα, πολύ ενθαρρυντικό, αν και αυτή τη στιγμή αναδιαρθρώνεται. Σε ό,τι αφορά το GSA, και την εφαρμογή του σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα μπορούσε να γίνει βάση της συνολικής διαχείρισης του προγράμματος. Γιατί το GSA θα είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται όλοι οι βασικοί παράγοντες για τη διαχείριση του προγράμματος. Ε, Από το 2014 στο 2015 πιστεύω ότι θα έχουμε εξασφαλίσει την, την πλήρη εφαρμογή του Γαλιλαίου. Θα είναι πλήρως επιχειρησιακό και λειτουργικό. Εγώ αυτό το χρονικό ορίζοντα δίνω 2014-2015. Και τότε θα γίνει μια σωστή αξιολόγηση των υπηρεσιών για να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε και στις εμπορικές υπηρεσίες. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι εταιρείες που είναι αρμόδιες για, την εφαρμογή, για τις εφαρμογές στις μεταφορές στις οδικές μεταφορές για παράδειγμα, πώς μπορούν ε, να, χρησιμοποιήσουν τις δικές μας οδηγίες. Πάντως υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές στον τομέα αυτό και μπορούμε να πούμε ποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ποιο τρόπο. Γιατί οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές χρησιμοποιούνται σε πολλές οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε έχουμε σημεία αναφοράς και για τις υπόλοιπες εφαρμογές. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Μπαρσιπατάκη ήθελε να πει δύο πράγματα ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια για τα εισοδήματα. Όπως ήδη ανέφερα, το σχέδιο δράσης ε, για την εφαρμογή πρέπει να επιταχυνθεί. Αλλά να σας ενημερώσω για τον κανονισμό 2008, ιδιαίτερα για την διαλειτουργικότητα του συστήματος. Νομίζω ότι το ζήτημα δεν έχει ακόμη επιληθεί. Το Κοινοβούλιο έχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ, γιατί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει την ε, κανονιστική διαδικασία του ελέγχου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιταχυνθεί η τυποποίηση. Χρειαζόμαστε την τυποποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που έχει το Κοινοβούλιο στα χέρια του για να επιταχύνει την εφαρμογή και συγκεκριμένα τα, τους πόρους, τα έσοδα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την Κομισιόν εάν συμφωνείτε. Κύριος Φερχεύ, μπορείτε να μας ε, πείτε ίσως κάποια και ακόμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ όλους τους ειδικού ε, του πάνελ για τις ε, συνεισφορές τους. Νομίζω πως αυτό το οποίο είδαμε είναι πως είναι τα ζητήματα του λέω πάρα πολλά, από ζητήματα διαχείρισης ε, έργου μέχρι νομικά, ρυθμιστικά, χρηματοδοτικές πτυχές, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Βεβαίω ε, δεν νομίζω ε, κανένα από τα ζητήματα αυτά δεν θα αυτό μιλήσουμε τα επόμενα χρόνια. Να πω λίγα πράγματα τώρα για την κάθε παρέμβαση και μετά να συνοψίσω με κάποιες γενικές σκέψεις. Πρώτα απ' όλα στην πρώτη παρουσίαση νομίζω τονίστηκε ο ρόλος ε, των ΜΜΕ. Βλέπετε και στην φάση των ε, προμηθειών καταβληθεί με προσπάθεια. Τώρα οι επιχειρήσει επιχειρήσεις στις υποδομές και στο διάστημα είναι κάτι πολύ περίπλοκο γιατί χρειάζεται πολύ, χρειάζονται πολύ εξειδικευμένες μικρομεσές επιχειρήσεις. Αλλά υπάρχει λόγος βεβαίω και για τις αγορές της, προς τα Κατάντη, προς την Λιανική και νομίζω πως εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία είναι βεβαίως ένας τομέας που απαιτεί μεγάλο μέγεθος επιχειρήσεων για να εμπλακεί αλλά, στο διάστημα γενικά, αλλά η δορυφορική πλοήγηση προσφέρεται και για μικρότερες επιχειρήσεις. Βεβαίως χρειάζεται οπωσδήποτε πείρα στον τομέα των μηχανικών κτλ. Αλλά και με λίγους ανθρώπους ήδη μπορεί να γίνει μια αρχή και αυτό είναι σημαντικό γιατί σημαίνει πως σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε όλα τα καρδιμέλη, σε όλες τις περιφερειές μπορούμε να έχουμε άμεσο όφελος για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίση σημαντική είναι η διάχυση της γνώσης. Αυτή τη στιγμή στείλουμε ένα νέο site, μια νέα ιστοσελίδα που θα τροφοδοτεί η Κομισιόν, και η GSA ω ε, μια κοινή πύλη πληροφόρηση. για τα τεχνικά δεδομένα για να γίνει πόρος για όσοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Όσον αφορά δε το ερώτημα της κυρίας Μπαρσιπατάκη, την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Σημαντικό είναι επίσης μετά από 10 χρόνια συζητήσεων για το ναι ή όχι ίσως ε, ε, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, υπάρχουν συμβάσεις, έχουμε και ημερομηνίες παραδοτέων Στι συμβάσεις. Είναι σημαντικό αυτό, δίνουμε σαφή μηνύματα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σοβαρή και βεβαίω μπορούν να γίνουν και οι απαραίτητες επενδύσεις ε, στον τομέα μετά των καταναλωτών της Λιανικής. Όπως είπαμε υπάρχουν πολλές προκλήσεις ε, μπροστά μας, να τονίσω μία. Ο ρόλος του ε, System On είναι κάτι το σημαντικό και καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εξαίρεση ορισμένων άλλων έργων. Είναι μια τελείως καινούρια διάσταση και προφανώς ε, πρέπει να υπάρξει και δημοσιονομική διαχείριση. Πρέπει δηλαδή να διαχειριστούμε σωστά αυτούς τους πόρους και για τον προπολογισμό και για το ίδιο το έργο. Έχουμε ήδη λοιπόν ξεκινήσει την εργασία από αυτού και θα επεκταθεί μέσω του προγραμματισμού στο μέλλον. Όσον αφορά την παρέμβαση του κ. Τορτόρα, νομίζω συμφωνούμε πως η δυνατότητα διαχείρισης του προγράμματος είναι πολύ σημαντική. Είναι κάτι το καινούργιο για την Κομισιόν υπό την έννοια πως ε, κατά βάση διαχείριση προγραμμάτων που κάνουμε αφορά την διαχείριση επιδοτήσεων εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά νομίζω πως αρκετά από αυτά τα οποία ανέφερε τα έχουμε ήδη κάνει. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι τι θα κάνουμε μακροπρόθεσμα και αν πράγματι είναι δουλειά της ε, Κομισιόν ή αν πρέπει να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. Όσον αφορά την παρα... παρουσίαση του κ. Τάρεκ για τις ε, εφαρμογές πρέπει να πούμε πως ε, οι εφαρμογές είναι ίσως ε, το πιο σημαντικό. Οπωσδήποτε η υποδομή είναι κάτω συναπαστικό, εκτοξεύουμε πυράβλους, ε, δορυφόρους, ε, κοστίζουν πολύ βεβαίως όλα αυτά, αλλά οι εφαρμογές της λιανικής είναι το σημαντικό και εδώ πέρα είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές. Δείχνουμε με τους υπολογισμούς μας πως η παγκόσμια αγορά για προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης και υπηρεσίες μέχρι το 2025 θα είναι γύρω στα 250 δισεκατομμύρια το έτος. Πάντα η ευρωπαϊκή βιομηχανία έλεγε πως θα πρέπει να καταλάβει το 1 τρίτο αυτής της αγοράς, δηλαδή μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια το έτος. Με το κόστος αυτού του συστήματος, και θα σας δώσω ένα νούμερο που ελέγχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά οι μελέτες δείχνουν πως ένα σύστημα αυτού του είδους Γαλιλαίο και Έγνος μαζί θα μας κοστίσουν γύρω στα 750 εκατομμύρια το έτος. Εάν ε, είναι αυτό το κλειδί για να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσουν τα συστήματα και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν αυτό αποτελέσει ένα καταλήτη ε, για να ανοίξει αυτή η αγορά των 70 δισεκατομμυρίων το έτος, νομίζουμε πως είναι μια καλή επένδυση. διστάζω λίγο για τις παρατηρήσεις ε, που έγιναν ε, για τις ε, αιτήσει και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Να θυμάστε πως το Γαλιλαίο είναι ένα παγκόσμιο σύστημα. Οπότε το τι θα ρυθμίσουμε εμείς αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι παραπέρα. Δηλαδή οποιαδήποτε υποχρεωτική χρήση μέσω κανονισμού του Γαλιλαίου μπορεί να λειτουργεί στην Ένωση αν αυτό θέλουμε. Αλλά δεν νομίζω να λειτουργεί στον υπόλοιπο κόσμο και το ζήτημα είναι μετά εάν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Π.χ. θα γίνει μια συμφωνία με την Ελβετία για να υπάγεται και εκεί χρήση στον ίδιο κανονισμό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να αναπτυχθούν ε, εφαρμογές και να μην υπάρχουν προβλήματα και εμπόδια και στην αγορά της Ένωσης, αλλά πρέπει να θυμόμαστε εδώ πως είναι ένα παγκόσμιο σύστημα. Επίσης, ετέθη το ερώτημα στις ε, περαιτέρω παρεμβάσεις ε, από τους βουλευτές ποιο είναι το πιο σημαντικό πολιτικό ερώτημα που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, το πιο σημαντικό πολιτικό ερώτημα είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει να δώσει μια μακροπρόθεσμη ε, δέσμευση. Γιατί αν δεν έχουν οι χρήστες αυτή την αίσθηση και πως θα υπάρχει μία ελάχιστη χρηματοδότηση, πως θα υπάρχει ένα παγκόσμιο μοντέλο διαχείρισης, τότε είναι απίθανο να επενδύσουν και να αναλάβουν τον κίνδυνο. Π.χ. εάν δούμε τον τομέα της αεροπορίας θα πρέπει να εξοπλίσουν με δέκτες ε, κάθε αεροσκάφος, πρέπει μετά να υπάρχουν διαδικασίες για τη χρήση τους ε, στα αεροδρόμια, πρέπει να πιστοποιηθεί ο εξοπλισμός, να εκπαιδευτούν οι πιλότοι, κοστίζουν πάρα πολύ όλα αυτά και ε, θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις εάν έχουν την εντύπωση και τις διαβεβαιώσεις πως και στις επόμενες και στις μεθεπόμενες δημοσιονομικές προοπτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματός της. Οπότε το ζήτημα δεν είναι τι θα κοστίσει και πώς θα το κάνουμε, αλλά εάν έχουμε την δυνατότητα να το υποστηρίξουμε γενικώ. Η γενναία απόφαση του 2008-2010 να ξεκινήσει η δημοπράτηση του συστήματος, ήταν αυτή, και το επόμενο ζήτημα το οποίο θα τεθεί σε λίγους μήνες είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί μια τέτοια παροχή πολυετή και πάνω σε αυτό να βασιστούν οι διάφοροι χρήστες, να χρησιμοποιήσουν τον καλαίο και το έγνος και να επενδύσουν στην χρήση των χρηστών της Λιανικής. Επίσης, οι Ρώσοι συναδελφοί έχουν υποφέρει ακριβώς από την έλλειψη τέτοιας δέσμευσης, οπότε περνάνε από κύκλους διαθεσιμότητας ε, της υποδομής που ανεβοκατεβαίνει, είναι, έχει διακυμάνσεις και έχει διακυμαθεί τρεις φορές ε, τελευταία και το γκλώνας άρα δεν υιοθετείται ε, εκτός Ρωσίας, ε, αν και η τελευταία δέσμευση ρωσικής κυβέρνησης είναι αρκετά σοβαρή. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε ποιο είναι το μελλοντικό μοντέλο σταθερής ε, διακυβέρνησης, πόσο κοστίζει και τι θα κάνουμε. Οι συζητήσεις αυτές είναι οπωσδήποτε πολύπλοκες. και αναμένουμε τις προτάσεις που αναφέρθηκαν με τη νέα Επιτροπή και τώρα θα φροντίσουμε να, να καταθέσει η Επιτροπή προτάσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να συζητηθούν στο δεύτερο εξάμεινο του έτους και μετά ελπίζουμε να έχουμε τον απαραίτητο κανονισμό και τους λοιπούς μηχανισμούς για να λειτουργήσει το σύστημα. Ε, θα ήθελα να μείνω σε αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τέλος να δώσω τον λόγο στον κύριο Ρέμεκ, τον εισηγητή μας ε, για να μας πει τη δική του αξιολόγηση και ίσως να μας πει τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Έχετε τον λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Είμαι ο εισηγητής υπεύθυνος για αυτήν την έκθεση, η οποία ονομάζεται έκθεση μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης, ενδιάμεσης αναθεώρησης, συγγνώμη. Μια και βρισκόμαστε στο πλαίσιο αυτής της μίνι ακρόασης, νομίζω ότι πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι οι ειδικοί αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας και μας εξέφρασαν τις απόψεις τους και την οπτική τους. Νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων σήμερα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι συνιστά έμπνευση για μας. Το πιστεύω αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σήμερα στην συζήτησή μας. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα, πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις και σχόλια ακούστηκαν σήμερα και όλα αυτά συμβάλλουν όχι μόνο στο ίδιο το σύστημα, αλλά και στην έκθεση της οποίας έχω την ευθύνη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η παρουσίαση του κύριου Μπενετό επιβεβαίωσε τις προσδοκίες μου, ιδίως όσο αφορά την ε, θέση των περιφερειών απέναντι στο Γαλιλαίο. Γιατί πιστεύω ότι το περιφερειακό επίπεδο είναι εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες μας και συνιστά το σύνδεσμο μεταξύ της Ευρώπης, το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να είναι εποφελές για τον καθένα από εμάς, για όλους τους πελάτες τους πολίτες μας. Επίσης εκτιμώ την παρουσία της κυρίας Μπάρση Πατάκη. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ειδική στον τομέα, είναι ειδική σε όλους τους τομείς της δορυφορικής πλοήγησης και των συναφών συστημάτων. Έχει έχει μια πάρα πολύ καλή στρατηγική και πολιτική ε, θέση ως προς τα οικονομικά και όλα τα άλλα ζητήματα των προγραμμάτων και θα χαρώ πάρα πολύ αν θα μπορέσουμε να εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε και την ευχαριστώ εκ βαθέων που δέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Τορτόρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας παρουσίαση. Πολλοί ανέφεραν ήδη τη σημασία της ποιοτικής διαχείρισης, της διαχείρισης της ποιότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος και όλοι το γνωρίζουμε. Προς τον κύριο Στάρεκ τώρα. Εκείνος ε, μας μίλησε για πολλές ε, εκφάνσεις, πολλά θέματα σχετικά με τα ωφέλη του προγράμματος Γαλιλαίος και, τον, και γενικότερα των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης. Ήταν όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα για όλους μας και για μένα ιδιαίτερα είναι σημαντικό ότι ο κύριος Στάρεκ εκπροσωπεί τη νέα γενιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η νέα γενιά βλέπει τον Γαλιλαίο ως ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμο, μακράς πνοής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα θα έχουμε άριστη συνεργασία στο μέλλον. Προσωπικά Είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζετε τις προσωπικές μου απόψεις, οπότε δεν θα τις εκθέσω αναλυτικά. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσετε να διαβάσετε πολλές από τις απόψεις μου και στην αιτιολογική έκθεση, η οποία θα υπάρχει στην ε, έκθεση αυτή, της οποίας φέρω την ευθύνη. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι Κάθε πρόγραμμα συνήθως έχει τρεις διαστάσεις, τρία θέματα, για να το πούμε απλουστευτικά. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα των οικονομικών. Το γεγονός ότι πολλά προγράμματα καθυστερούν, ε, γιατί είναι ανταγωνιστές στο παγκόσμιο επίπεδο. Φέτος υπάρχουν 62 και τα τελευταία 40 χρόνια συμμετείχα σε πάρα πολλά διαφορετικά προγράμματα, διαφορετική σημασία σίγουρα, αλλά κανένα από αυτά τα προγράμματα δεν αντιμετωπίστηκε διαφορετικά. Το, όλα τα προγράμματα, το κάθε έδωσε τη δική του μάχη για τα οικονομικά, για την έλλειψη πόρων. Σίγουρα υπάρχει πολύ σφοδρός ανταγωνισμός μεταξύ των προγραμμάτων. Προσωπικά πιστεύω ότι θα υπερβούμε όλα αυτά τα προβλήματα και τις δυσκολίες και θα εκτιμήσετε το γεγονός ότι ε, καταφέραμε και χρονικά να εντάξουμε αυτή την ακρόαση στη διαδικασία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω τις απόψεις σας με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ και εγώ για την καλή σας ε, προετοιμασία, για την συνεισφορά και είμαι σίγουρος ε, πως θα τα συζητήσουμε και τα συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα εντατικά, ακούσαμε και τους συναδέλφους και βεβαίω μετά θα ληφθεί μια απόφαση. Για σήμερα όμως τελειώσαμε, οπότε σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά και τον κύριο Ρέμεκ και τους εμπειρογνώμονες και εδώ πέρα τελειώνει η συνεδρίασή μας. Να σας παρακαλέσω οι υπάλληλοι της ομάδας να φέρουν τους συντονιστές ε, λίγο πιο σύντομα μέσα για να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Ευχαριστώ.